Ε, κυρία Μάισνερ, κυρίες και κύριοι, ακόμα παραμένουν πολλοί στην αίθουσα. Θα φανταστικό. Μη φοβηθείτε ότι θα υπάρξει άλλο πάνελ που θα μακρηγορήσει. Απλώς τα καταληκτικά σχόλια και θα δώσω το λόγο στον Επίτροπο Βέλα να κάνει τις θεματικές ε, ε, καταληκτικές παρατηρήσεις και εγώ τις ευχαριστίες για να κηρύξουμε το πέρας αυτής της διοργάνωσης. Ευχαριστώ πολύ Γκεζινέ, αξιότιμα μέλη, κυρίες και κύριοι. Καταρχάς θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για αυτό το απόγευμα. Μεγάλη πηγή έμπνευση οι παρουσιάσεις και πολύ ενδιαφέρουσα ήταν η συζήτηση. Και πολύ ενθαρρυντικό είναι να βλέπουμε ότι όποιε και αν είναι οι προτάσεις μας, οι πολιτικές μας απόψεις, συμφωνούμε όλοι για το εξή ότι χρειαζόμαστε μια δράση ισχυρή και συντονισμένη για τον κανονισμό, για τον, τους ωκεανούς μας, συγγνώμη. Αλλιώς η οικονομία μας κινδυνεύει και οι ζωές μας οι ίδιες και το περιβάλλον. Τα τελευταία χρόνια η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει αναλάβει πολύ φιλόδοξη δράση για να μειώσει την παραγωγή πλαστικών, να καταπολεμήσει τη λαθρέα αλληλεία και να καταστήσει τα αποθέματα βιώσιμα, έτσι ώστε να υποστηρίξει την γαλάζια οικονομία να αναπτύξει τη θαλάσσια έρευνα και την επιτήρηση των ωκεανών. Όπως γνωρίζετε, παραμένουν μεγάλες όμως οι προκλήσεις. Τα ωκεάνια συστήματα είναι περίπλοκα και είναι πολλές οι πιέσεις, κλιματική αλλαγή, ρήπανση, βιοπικιλότητα και απώλειά της και υπεραλίευση. Όλα αυτά θα εξακολουθήσουν να ε, ε, πλήττουν τους ωκεανούς. Μέχρι το 2050 θα είμαστε 9 με 10 δισεκατομμύρια άνθρωποι στη γη και θα αυξηθούν οι πιέσεις όλες αυτές. Θέλω να σας ε, ε, διαβεβαιώσω ότι είναι προσιλωμένη σε αυτή την προσπάθεια πλήρωση η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να υποστηρίξει τις δράσεις είτε πρόκειται για το νέο πρόγραμμα Horizon ε, Europe ε, εστίαση στους ωκεανούς, είτε ε, στη νέα θαλάσσια στρατηγική και το Ταμείο μετά το 2020 για τη θάλασσα και την αλία. Και επίσης για την εξωτερική χρηματοδότηση και το αντίστοιχο μέσο μετά το 2020. Είναι παγκόσμιο ηγέτης, αξιόπιστος η Ευρωπαϊκή Ένωση και είναι προσιλωμένη και παραμένει στο να πρωταγωνιστεί διεθνώς στα πλαίσια των Ηνωμένων Εθνών, τη ατζέντα του 2030 για τη βιώσιμη ανάπτυξη και στην εφαρμογή της συνθήκης του Παρισιού, της συμφωνίας μάλλον, και για την προστασία της θαλάσσιας βιοπικιλότητας στις ανοιχτές θάλασσες και τους ωκεανούς. Και ξέρουμε ότι για να παραμείνουν υγιείς οι ωκεανοί θα πρέπει όλοι μας να συνεργαστούμε στενότερα. Για το λόγο αυτό και μαζί με τη συνάδελφό μου Γκερίνη χαράσουμε ένα φόρουμ για τη διακυβέρνηση των ωκεανών παγκοσμίω, με εμπειρογνώμονε, με εκπροσώπου κοινωνία των πολιτών, πανεπιστημιακού ερευνητέ και ε, ανθρώπους που λαμβάνουν αποφάσεις για να δώσουν συνέχεια στις δικές μας προτεραιότητες, για να συζητήσουμε τις διεθνείς προκλήσεις και προβλήματα και πιο σημαντικό για να συστήσουμε δράση. Αυτό θα είναι ένα ακόμα βήμα στις προσπάθειές μας για μια πιο ολοκληρωμένη προσέγγιση ε, προς τους ευρωπαϊκούς και παγκόσμιους Οκεανούς. Θα μπορούσε να δημιουργηθεί και μια επιτροπή ωκεανών στο επόμενο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, μια μόνιμη επιτροπή. Και χρειάζεται και περαιτέρω δράση. Φυσικά θα συνεχίσουμε στο δρόμο αυτό και ελπίζω και εσείς να συνεχίσετε και να συναντηθούμε για να συνεργαστούμε για ένα καλύτερο γαλάζιο ωκεανό. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Thank you very much, Ευχαριστώ πολύ, Καρμενουβέλα. Χαίρομαι πάρα πολύ που παραμείνατε μέχρι το τέλος. Καλά και εγώ παρέμεινα. Αλλά Ήθελα να γίνει αυτή η διάσκεψη εδώ και πάρα πολύ καιρό και φυσικά θα παραμείνω, αλλά ε, συνήθω οι επίτροποι έχουν τόσε πολλέ υποχρεώσει και αντισταθήκατε σε όλου του πειρασμού και παραμείνατε εδώ. Είναι θαυμάσιο αυτό και πραγματικά ένα ε, προσεκτικός παρατηρητής καταλαβαίνει ότι τα λαμβάνετε αυτά σοβαρά υπόψη και το ξέρω εγώ φυσικά ότι τα λαμβάνετε σοβαρά υπόψη. Λοιπόν, πρέπει να σας κάνω ένα σχόλιο επειδή είπα ότι ορισμένοι ρωτούσαν γιατί έχει πλαστικό καπάκι αυτό το μπουκάλι. Έχει μια ιστορία το μπουκάλι αυτό. Συνήθως εδώ έχουμε παντού πλαστικά μπουκάλια. Και ε, ε, το δικό μας Intergroup ε, αρνήθηκε να έχει. Έχει μόνο ποτήρια και γυαλί. Αυτό είναι ένα συνδυασμό από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Το καπάκι είναι πλαστικό, αλλά είναι ανακυκλούμενο. Το άλλο είναι γυαλί. Και το κοπάνισα. Πάντως θα πρέπει να ε, σκεφτούμε πώς ε, να ε, αποφύγουμε να έχουμε μπουκάλια πλαστικά μιας χρήσης. θέλω να πω και άλλα. Ήταν συναρπαστική αυτή η διάσκεψη. Ικανοποιήθηκα πάρα πολύ και είμαι πανευτυχής που το καταφέραμε να συγκεντρώσουμε τόσο κόσμο. Ε, ε, χίλιοι εγγεγραμμένοι είναι πολύ. Εγώ θα προτιμούσα ένα εκατομμύριο. Θα ήταν ακόμα καλύτερα. Ε, να γνωρίζει ένα εκατομμύριο κόσμο τι γίνεται με τους ωκεανούς είναι μια καλή αρχή πάντως και η χίλιοι. Και ως ε, ιδέα είναι θαυμάσια και λαμπρή ιδέα ε, για ε, έναν οργανισμό για τους ωκεανούς εκτός από τη Γενική Διεύθυνση ΜΑΡΕ. Και τώρα έχω τη χαρά και την ευχαρίστηση να σας ευχαριστήσω όλους. Όλους τους προσκεκλημένους, τους γιατί χωρί κοινό δεν θα μπορούσαμε να έχουμε διάσκεψη. Ευχαριστώ όλου του συναδέλφου, ομιλητέ, ομιλητέ από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Εγώ ποτέ δεν έχω δει διάσκεψη με υψηλού επίπεδου με τόσου πολλού ευρωβουλευτέ. Έτσι δεν είναι πολύ μεγάλη επιτυχία γιατί θα πρέπει να έχουμε ένα πολλαπλασιαστικό ρόλο. Ευχαριστώ όλου όσοι διοργάνωσαν, ιδιαίτερα το ιδιαίτερο γραφείο ε, του Προέδρου Ταγιάννη και κυρίως την κυρία Μαγδαλένα Πιόρουν και Γκοσάλη Μεντόσα Ασένση, αλλά κυρίως τη Γενική Διεύθυνση Μάρε, Ραμόν Βαν Βάλτεβελ και την Αλεξάνδρα Λαμόρ που είχαν πολλή δουλειά και εκτός αυτού θα ήθελα και πάλι να αναφέρω γιατί ξέχασα μια γενική διεύθυνση στα εισαγωγικά μου σχόλια Γενική Διεύθυνση Director, Director General είναι στα αγγλικά ΜΑΡΕ και RTD, αλλά και περιβάλλοντος. Ε, ε, ξέχασα να την αναφέρω αυτή τη Γενική Διεύθυνση Περιβάλλοντος Ευρωπαϊκής Επιτροπής, που είναι επίσης πάρα πολύ σημαντική. Και τώρα, χωρίς αυτό να είναι το λιγότερο σημαντικό, ένα τελευταίο. Όλοι εσείς εδώ παρόντες αγαπάτε τους ωκεανούς. Για μένα είναι κρίσιμο να βλέπουμε ότι χρειάζεται προστασία ωκεανός. Ε, ένα πλανήτη έχουμε μόνο. Αυτό το πλανήτη έχουμε, αυτούς τους ωκεανούς. Πρέπει να τους προστατεύουμε. Και ο κόσμος προστατεύει ό,τι αγαπάει. Λοιπόν, φεύγοντας από εδώ θα πρέπει όλοι να προσπαθήσουμε να βγούμε και να κάνουμε τους άλλους ανθρώπους να αγαπήσουν τους ωκεανούς. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθατε.